Πρώτα, μία ανακοίνωση. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος στην έναρξη της Συνόδου, οι κύριοι Μπονάνο και Μίκη έχουν ένα αίτημα. Πρόκειται για κυρώσεις που θα επιβληθούν στους δύο αυτούς